τους συναδέλφους για τις υπογραφές τους. Χάρη σε αυτούς το θέμα των αδέσποτων σκύλων μπορεί να βρει μια λύση. Ε, Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζουμε και παίρνουμε στις ψηφοφορίες. Το πρώτο θέμα είναι η έκθεση ε, του κυρίου Ρικέ Ε, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είναι η συμφωνία με το Πράσινο Ακροτήριο για ορισμένε πτυχέ αερομεταφορών. Το επόμενο θέμα που θα ψηφίσουμε είναι τα συστήματα εγγύηση ασφαλίσεων του κυρίου Σκίνερ. Έκθεση ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Επόμενη έκθεση του κυρίου Κάζα το μέλλον του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το λόγο έχει ο εισηγητής για προφορική τροπολογία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παράγραφος 13 καλύπτεται εν ε, από ένα τμήμα της ΕΝΕΑ και για να μην έχουμε απικαλύψεις ε, ζητώ με προφορική τροπολογία να απαλληφθεί η παράγραφος 13. Έχω δε πληροφορηθεί ότι συμφωνούν και άλλες πολιτικές ομάδες με την προφορική αυτή τροπολογία. Ο Πρόεδρος. Διαφωνεί κανείς με την προφορική τροπολογία του κυρίου Κάζα. Παρακαλώ να γερθείτε αν διαφωνείτε. Όχι. Δεν βλέπω αντιρρήσει. Ψηφίζουμε λοιπόν το κείμενο της εκθέσεως όπως τροποποιήθηκε με την προφορική αυτή τροπολογία και ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ευχαριστούμε κύριε Κάσα. Επόμενο θέμα σήμερα μέση διάταξη. Η έκθεση της κυρίας Μπόουλς για το διορισμό ενός ε, μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρόκειται για τον κύριο Άσμουσεν. Μυστική ψηφοφορία. Παρακαλώ, θα χρησιμοποιήσουμε τα μηχανήματά μας και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το φως που θα δείτε στα μηχανήματα θα είναι μπλε και κανένα άλλο χρώμα. Μόλις ψηφίσετε, επειδή είναι μυστική ψηφοφορία δεν θα δείτε άλλα χρώματα παρά μόνο ένα μπλε φως. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Προς το νέο μέλος. Και ευχαριστούμε την κυρία Μπόλς για την έκθεσή της. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με κάποιο μηχάνημα που δεν λειτουργεί θα στείλουμε τεχνικό. Επόμενο θέμα. Εγγραφή για την απόκτηση νέων μεριδίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Όχι, δεν είναι αυτή ζητώ συγγνώμη, είναι η έκθεση του κυρίου Κάλφιν, χορήγηση εγγύηση Ευρωπαϊκή ε, Ένωση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χωρί τροπολογίε. Ούτε πρόταση απόρριψη ε, έχω, οπότε εγκρίνεται η κοινή θέση του Συμβουλίου. Τώρα ε, ακολουθεί η έκθεση Τη κύρια Μπόλς που σα είπα προηγουμένω εγγραφή για την απόκτηση νέων μεριδίων στο μετοχικό κεφάλαιο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζας για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Ω αποτέλεσμα ε, τη απόφαση αύξηση ε, κεφαλαίου ψηφίζουμε ψήφι υπέρ του μπλοκ υπαριθμών 1 κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε ψηφιπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια κυρία Μπόουλς. Επόμενη έκθεση. Εφαρμογή του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα και θέσπιση άδεια εξαγωγή καθώ και μέτρων εισαγωγή και διαμετακόμιση για πυροβόλα όπλα, μέρη και εξαρτήματά του και πυρομαχικά. Είναι έκθεση του κυρίου Γιακολίνο που θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Πολύ σύντομη παρέμβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, του κλάδου. Σημαίνει αυτό απλούστευση, λιγότερο κόστος, λιγότερο διοικητικό άχθος και γραφειοκρατία, σαφή μέτρα και συγκεκριμένα για την εξαγωγή πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτική χρήση, καταπολέμηση του λαθρεμπορίου όπλων και καλύτερη χνηλασιμότητα των όπλων που κυκλοφορούν και μάλιστα σε ένα σύστημα το οποίο συνεχώς διευρύνεται. Είναι η πρώτη συγκεκριμένη απάντηση στις τραγικές ε, εξελίξεις και τραγικά γεγονότα που γνωρίσαμε στην Ορβηγία. Αυτό αφορά πολλούς ενεχομένους στον κλάδο που ε, ασχολούνται ε, με τα όπλα ε, ως άθλημα. Ευχαριστώ. Και τώρα ψηφίζουμε συμβαστική τροπολογία υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σχέδιο προτάσεως Επιτροπής υπέρ παρακαλώ όπως τροπήθηκε κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε. Τώρα την ε, πρόταση με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια μου στον συγκεκριμένο. Η επόμενη έκθεση είναι του κυρίου Μορέιρα. Εξαιρετικά εμπορικά μέτρα για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά αποχές. Έγκρινεται. Η πρόταση πώς τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα παρακαλώ με ονομαστική ψηφοφορία. Τώρα άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Το επόμενο θέμα για τη διάταξη είναι τρεις προτάσεις ψηφίσματος σχετικές με την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχέδιο ψηφίσματος υπαριθμών. Σχέδιο ψηφίσματος τεσσάρων πολιτικών ομάδων. Έχουμε τμήματα στην τρίτη παράγραφο. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Στο 5. Σημείο 2, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 5 πάντα. Σημείο 4, παύλα 4, δύο τμήματα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Παύλα 5. Πρώτο τμήμα. χωριστή ψηφοφορία μόνο, δεν υπάρχει το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5, Παύλα, ε, υπαριθμών 5 εγκρίνεται και περνάμε στην Παύλα υπαριθμών 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το σύνολο της προτάσεως ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ως εκ τούτου οι λοιπές προτάσεις ψηφίσματος καταπίπτουν και έχουμε το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, δύο προτάσεις ψηφίσματος για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σέγγεν. πρόταση ψηφίσματος των πέντε πολιτικών ομάδων με την τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο της προτάσεως ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και έτσι ολοκληρώνω την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ.